νομίζω ότι θα είμαστε μια πιο ε, θα έχουμε πιο στενές σχέσεις με όλους τους εταίρους στο εξωτερικό εμπόριο. Ευχαριστούμε Βίταλ. Κλείνει η συζήτηση και η ψηφοφορία θα λάβει η χώρα αύριο στις 12 το μεσημέρι. Στη συνέχεια έχουμε άλλη μια έκθεση του Βιτάλ Μορέιρα μακροοικονομική χρηματοδοτική σύνδρομη στην Δημοκρατία της Κυργιζίας. Έχετε το λόγο, ε, κύριε Μορέιρα. Γνωρίζετε ότι έχετε στη διάθεσή σας έξι λεπτά, τέσσερα τώρα και δύο για να κλείσετε. Αλλά μπορείτε να κάνετε του χρή... χρήση του χρόνου σας όπως επιθυμείτε. Δυστυχώς δεν έχω ιδιαίτερα καλά νέα. Εγώ εκπροσωπώ τη θέση της Επιτροπής ε, Διεθνούς Εμπορίου και υπάρχει μεγάλη ε, ρήξη με το Συμβούλιο. Η Ίντα λοιπόν προτείνει μία πρόταση της Κομισιόν του Δεκεμβρίου 2011 για μακροοικονομική αρρωγή προς τη δημοκρατία της Κυριζίας ε, της τάξης του, των 30 εκατομμυρίων ευρώ έγινε και μία μικρή τροποποίηση έτσι ώστε να αλλάξει η συμβουλευτική διαδικασία, η διαδικασία διαβούλευσης ως προς την ε, επιτροπολογία δηλαδή για την εκτέλεση της συμφωνίας. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να φτάσουμε σε συμφωνία με το Συμβούλιο επί του θέματος. Η ίντα υποστήριξε ότι χρειάζεται η διαδικασία επιτροπολογίας, κάτι το οποίο μπορεί να αφιερζητηθεί. Τα διάφορα ε, μνημόνια θα πρέπει να εγκριθούν με βάση διαδικασία διαβούλευσης, όπως ίσχυε με τη, ίσχυσε με τη Μολδαβία και την Ουκρανία. Και θα πρέπει τα κράτη-μέλη να έχουν τη δυνατότητα να προβάλλουν δικαίωμα άρνηση κυρίας ως προς τις εξουσίες της Κομισιόν. Το Συμβούλιο θεωρεί ότι η διαδικασία διαβούλευσης θα πρέπει να είναι μια έκτακτη διαδικασία μετά από υποστήριξη αναπερίπτωση. Όμως το Συμβούλιο άλλαξε θέση στο μεταξύ διότι Γίνεται λόγος για, δηλαδή μάλλον βασίστηκε στις μακροοικονομικές συμφωνίες με την Ουκρανία και τη Μολδαβία. Το μήλο της έριδος δεν αφορά θέμα ουσίας. Υποστηρίζουμε την αρρωγή αυτή προς το Κυργιστάν. Υπάρχουν δύο αλληλένδετα πολιτικά ζητήματα. Ένα θεσμικό για να δούμε ποιος είναι ο βαθμός ελέγχου που διαθέτουν τα κράτη-μέλη με βάση τις εκτελεστικές εξουσίες της Επιτροπής και υπάρχει και ένα άλλο θέμα που έγκυται στο εξής. Το Κοινοβούλιο μπορεί να δεχτεί ενισχυμένο έλεγχο του Συμβουλίου διαμέσου των κρατών μελών τη στιγμή που το Κοινοβούλιο δεν μπορεί να ελέγξει κατά παρόμοιο τρόπο την Κομισιόν. Γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε στεναρή θέση ως προς την ισορροπία αρμοδιοτήτων που ορίζει η συνθήκη της Λισαβόνας και δεν δεχόμαστε τις μηχανοραφίες του Συμβουλίου μέσω επιτροπολογίας για να μην υπάρχει ίση κατανομή αρμοδιοτήτων. Αυτή η στρατηγική δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Δεν μπορεί το Συμβούλιο να ακολουθεί ερετική θέση διακυβεύοντας τα δικαιώματα της ε, Κυργιζίας, της Ουκρανίας και της Γεωργίας. Ο Επίτροπος έχει το λόγο για να μας πει τη θέση της Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Θα ήθελα ξεκινώντας να σας πω ότι η μακροοικονομική βοήθεια της Ένωσης είναι σημαντικό μέσο για τις σχέση με τις γειτονικέ και υποψηφίες χώρες. Λόγω των αρνητικών επιπτώσεων της ε, ε, κρίσης στην περιοχή μας, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συμπληρώσει τις προσπάθειες του ΔΕΛΤΑΝΙΤΑΦ για την στήριξη των ε, περιοχών των χωρών αυτών. Αυτή τη στιγμή η μακροοικονομική βοήθεια δεν προωθείται. Μετά από τις προτάσεις της Επιτροπής για τη Γεωργία του Ιανουαρίου 2011, τα Κοινοβούλια και το Συμβούλιο διαφώνησαν στη χρήση της διαδικασίας της Επιτροπολογίας, όπως πολύ σωστά τόνισε και ο καθηγητής Μορέλα. Η Επιτροπή πιστεύει ότι προέχει να βρούμε μια λύση στα πλαίσια μιας εξεταστικής διαδικασίας για την εφαρμογή του Μνημονίου Συναντήληψης. Για την περίπτωση της Γεωργίας και του Κυρικιστάν, οι μακριές καθυστερήσεις στη λήψη αποφάσεων έχουν, έχουν θέσει σε δύσκολη θέση την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, Φαίνεται ότι το πρόβλημα αυτό μπορεί να εμποδίσει την υποβολή συγκεκριμένων προτάσεων και αυτό θα έχει επιπτώσεις στη σχέση με την Αίγυπτο, την Ινσία και την Αρμενία που έχουν υποβάλει, πρόκειται να υποβάλουν αίτηση για τέτοια στήριξη. Καλή λοιπόν η Επιτροπή την, ε, ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να καταβάλει κάθε δυνατές προσπάθειες για να ξεπεραστεί το αδιέξοδο και να είναι πλέον διαθέσιμα τα μακροοικονομικά μέσα. η χορήγηση δηλαδή μακροοικονομικής χρηματοδυτικής συνδρομής και ελπίζουμε ότι θα υποβληθεί τη σχετική πρόταση στο Συμβούλιο. Είναι σημαντικό, όπως τον είχε καθεί Μορέλα, να εφαρμοστεί η συνθήκη της Λισαβόνας με την τήρηση όχι μόνο του γράμματος αλλά και του πνεύματος της Συμφωνίας της Λισαβόνας δεν μπορούμε να αντιληφθούμε γιατί μετά από τρία χρόνια δεν είναι δυνατόν να καταλήξουμε σε μια συμφωνία για ένα τόσο ευαίσθητο θέμα. Ε, μιλάμε για ένα σημαντικό πολιτικό εργαλείο για τις Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις γειτονικές χώρες, σε ό,τι αφορά τις σχέσεις με τις γειτονικές χώρες. Θα αρχίσουμε με τον γύρο των παρεμβάσεων εξ των πολιτικών ομάδων. Εξ ονόματος του ΕΛΚ και για δύο λεπτά το λόγο έχει ο κύριος Μπαρτολότσι. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η σημερινή συζήτηση για την ε, χρηματοοικονομική συνδρομή στο Κυργιστάν μας οδηγεί να δούμε πώς εξελίχθηκε η, κατάσταση, η πολιτική κατάσταση στη χώρα έτσι ώστε να επιτευχθεί μια σταθερότητα. Σήμερα βλέπουμε ότι υπάρχει μια σταθεροποίηση και σταθερότητα και οι συνταγματικές μεταρρυθμίσεις καθώς και οι προεδρικές εκλογές οδήγησαν στις μεταρρυθμίσεις που είναι αναγκαίες για να μπορέσει η χώρα να ανταποκριθεί στα δημοκρατικά δεδομένα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπάθησε να παρακολουθήσει την εξελικτική αυτή πορεία και προέβαλε σύνδρομη έτσι ώστε να στηρίξει έμπρακτα τη χώρα αυτή μέσα στα πλαίσια των δημοκρατικών και κοινωνικών μεταρρυθμίσεων. Γι' αυτό ελπίζω το νομικό ζήτημα που παραμένει ανοιχτό μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων που δεν επέτρεψε την ε, ψηφοφορία σε πρώτη, μετά από πρώτη ανάγνωση να μπορέσει να αντιμετωπιστεί έτσι ώστε να χορηγηθεί αυτή η σύνδρομη. Αυτές οι καθυστερήσεις επιπλέον ε, πέρα από το γεγονός ότι έχουν επιπτώσεις επί της χώρας επιβάλλουν και λειτουργούν αρνητικά ως προς την αξιοπιστία, τη διεθνή αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόσφατα ως αντιπροσωπεία μεταβήκαμε Μεταβήκαμε στο Κυργιστάν, Είναι, είμαι πρόεδρος της Μικτής Επιτροπής και είδαμε ότι από πλευράς αυτής της χώρας υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση σε σχέση με τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί. Ελπίζω το θέμα αυτό να επιληθεί έτσι ώστε να είμαστε πλέον αξιόπιστοι θεσμικά και να εγγυηθούμε την σταθερότητα και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας που είναι ζωτικής σημασίας για τη διεθνή ασφάλεια. Ευχαριστούμε κύριε Μπαρτολότσι. Εξ ονόματος των σοσιαλιστών και για 1,5 λεπτό ο κύριος Κούτας έχει το λόγο. Ευχαριστώ ε, πρόεδρε. Θα ήθελα Χαιρετίζω. να ευχαριστήσω για την ε, άμεση βοήθεια προς το Κυργιστάν το 30 εκατομμυρίων έτσι ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει τα άμεσα οικονομικά προβλήματα και προβλήματα των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Η εγκληματικότητα, η τρομοκρατία ε, ενυπάρχουν στη χώρα, γι' αυτό θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι οι εκλογές του 2010 οδήγησαν σε, μια, σε κλειδονισμούς και σε σειράξεις μεταξύ δύο μεγάλων εθνικών, δύο μεγάλων εθνοτήτων. Και γι' αυτό είπαμε ότι θα πρέπει να προωθήσουμε τη συμφωνία μεταξύ Δημοκρατίας του Κυργιστάν και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πέρα από το ε, νομικό ζήτημα, ελπίζω η Ευρωπαϊκή Δημοκρα... Ε, Διπλωματία να μπορέσει να διαδραματίσει σωστό ρόλο για να βοηθήσουμε αυτή τη δημοκρατία της Κεντρικής Ασίας. Ο κύριος Κάζαξιτ σε τον λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Βεβαίως η Κυρκυζία δεν βρίσκεται εντό του γεωγραφικού εύρους της ε, συμφωνίας αυτής, ε, αλλά Φαίνεται πως ε, έχει γίνει χάρη στις ε, μεταρρυθμίσεις οποίες προωθούμε ένα σημαντικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ε, περιοχή μέσω της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής βοήθειας η οποία φτάνει το ύψος των 30 εκατομμυρίων ευρώ. Βεβαίως υπάρχουν φόβοι για την διαχείριση ε, αλλά και για την ε, ασφάλεια των συστημάτων πληροφορικής, ε, της εσωτερικής συμμόρφωσης, για τα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων επίσης, αφότου ξέσπασαν εθνοτικές συγκρούσεις. Αλλά θεωρούμε πως η Κυργιζία, από ό,τι φαίνεται, κάνει κάποια βήματα προς σωστή κατεύθυνση και αν γίνει αυτό θα στείλει το μήνυμα στις άλλες χώρες περιοχής πως είναι σαφώς ε, ε, προς έναν δρόμο εκδημοκρατισμού. Παρ' αυτά, η Κομισιόν, εάν δεν υπάρξει πρόοδος, δεν θα πρέπει να διστάσει να αναστείλει τις πληρωμές της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής ε, περισσότερα για περισσότερα, αλλά και την αντίστροφη αρχή, λιγότερα για λιγότερα. Τώρα, όσον αφορά το βασικό ζήτημα του κυρίου, της έκθεσης του κυρίου Μορέρα για τη Συμφωνία Πλαίσιο για την Μακροοικονομική Χρηματοδοτική Συνδρομή στην Δημοκρατία της ε, Κυργιζίας. Συμβούλιο και Κοινοβούλιο πρέπει εδώ πέρα να δώσουν το παράδειγμα, να χρησιμοποιήσουν την κοινή λογική, να καταλήξουν σε μια λογική συμφωνία για να εφαρμοστεί η συνθήκη της Λισαβόνας. Σας ευχαριστούμε κύριε συνάδελφο. Κύριε συνάδελφε, η κυρία Κιλ Νίλσεν έχει το λόγο. Πρόεδρε, μετά τις ε, εθνικές σειράξεις στη χώρα και το ψήφισμα του νέου συντάγματος οδηγείται η χώρα προς τον εκδημοκρατισμό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστήριξε αυτή τη φτωχή χώρα που έχει πληγεί από την οικονομική κρίση. Το Κυργιστάν είχε επιλεγεί ως χώρα πιλότος για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Υποστήριξης στη Δημοκρατία τότε όμως έχει επιδεινωθεί η κατάσταση. Υπάρχουν στοιχεία για βασανιστήρια στα, στις φυλακές. Ο Ασταρόφ, ο οποίος ήταν υπεραξής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 61 ετών, ε, ε, είναι ουσβέκικης καταγωγής, ο οποίος ε, βρίσκεται διαβίου στη φυλακή. Δεν υπάρχει δυνατότητα να διατηρηθεί η σταθερότητα και η ηρεμία στη χώρα, δεν υπάρχει δυνατότητα συμφιλίωσης, ο εθνικισμός και ο ρατσισμός επιδεινώνονται, το κοινοβούλιο στην πρωτεύουσα ε, ε, ε, έγιναν επιθέσεις σε τρεις αδελφούς ουσμπέκικης καταγωγής και τέλη Νοεμβρίου ένας ερευνητής στην ελήφθη από το, τις, πράκτορες του τοπικού KGB, της τοπικής KGB οι πολλοί υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, ε, μόνο για το λόγο επειδή είχε ζητήσει να πάρει συνεντεύξεις από υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κυρία Άστον, η οποία μετέβη στο Κυργιστάν πριν από λίγο καιρό, δεν πήρε θέση ούτε για την καταδίκη του Ασκάροφ, ούτε για την παρενόχληση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν μπορεί να ε, συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Δεν μπορεί να δίνει τυφλά η χρηματοοικονομική συνδρομή, μακροοικονομική συνδρομή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να θέσουμε όρους απέναντι στην δημοκρατία αυτή, περιμένοντας σημαντικές προόδους σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της δικαιοσύνης και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Πάσκα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πάσκα. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, τα οικονομικά προβλήματα που προκάλεσε η κρίση του 2009 έχουν οδηγήσει σε μια εξέγερση στην Κυργιζία, την οποία ακολούθησε και εθνοτική βία. Η προσωρινή κυβέρνηση κατάφερε να σταθεροποιήσει την κατάσταση, να εφαρμόσει δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις και να οδηγήσει τη χώρα σε δημοκρατικές εκλογές. Όμως η εύθραυστη αυτή διαδικασία εξακολουθεί να απειλείται από την οικονομική αστάθεια και σύμφωνα με την ανάλυση του Δουνουτού η χώρα θα χρειαστεί να καλύψει ένα έλλειμμα 330 εκατομμυρίων ευρώ το 2011 και 2012. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει πως θα πρέπει να συνεχίσουμε την μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στη Δημοκρατία της Κυριγησίας μέσω δανείων και επιχορηγήσεων σε ποσοστό 50 και 50%. Εάν επαληθευτούν λοιπόν οι ειδικοί ότι δηλαδή η βοήθεια αυτή θα βοηθήσει τη χώρα να ξεπεράσει αυτή την κρίσιμη περίοδο και να οδηγηθεί σε σταθερότητα και στον τομέα των πολιτικών και των συγκρεώσεων και της δημοκρατίας, τότε θα ε, επιτύχει αυτή η βοήθεια του στόχου της. Μακροπρόθεσμα όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί το εάν τα κονδύλια αυτά έχουν το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Δίνω και καλωσορίζω τον ε, κύριο Μπόρκ, τον κύριο Επίτροπο που μόλις ήρθε. Η κυρία Στάσεν Λοάνς έχει το λόγο τώρα. Κύριε Πρόεδρε, η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια τεράστια οικονομική κρίση οι πολίτες τις γονατίζουν. Πώς είναι λοιπόν δυνατόν να γράφουμε επιταγές σε χώρες που απέχουν χιλιάδες χιλιόμετρα από εδώ πέρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να συμμαζέψει τα δικά της. Γιατί κάνει τέτοια πράγματα. Ε, από όταν ξεκίνησε η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή έχουν δοθεί γύρω στα 7 δισεκατομμύρια. Τα περισσότερα από αυτά δίνονται ως δώρο σε χώρες που έχουν γνωστή φήμη οργανωμένης εγκληματικότητας και διαφθοράς. Αυτή τη φορά λαμβάνει χρήματα η Κυργυζία. Μα η μακροοικονομική ε, συνδρομή πηγαίνει υποτίθεται σε χώρες γειτονικές. Η Κυργυζία είναι στην κεντρική Ασία, 6.000 χιλιόμετρα από εδώ. Απέχει όσο και η Κίνα. Πού θα σταματήσει αυτή η πρακτική. Παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα εκεί πέρα, συλλαμβάνονται ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι μία από τις πιο διεφθαρμένες χώρες στον κόσμο. Και δίνουμε 30 εκατομμύρια, από τα οποία τα 15 είναι δώρο. Ε. Βλέπουμε την ε, αντίθεση με την κατάσταση στην Ευρώπη. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή σκοντάφτει οικονομικά και κοινωνικά, αλλά παριστάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Και πληρώνει ο φορολογούμενος γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να κάνει τέτοια δωράκια στην Κυργιζή. Κύριε Πρόεδρε, πρόκειται πραγματικά για μια πολιτική τραγική. Πρέπει να σταματήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Τον λόγο έχει η κυρία Γέγκλε. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, καλώς ήρθατε. Εγώ είμαι υπέρ της ε, μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής ε, στην δημοκρατία της ε, ε, Αυτή τη στιγμή η χώρα βρίσκεται σε μια φάση σταθεροποίησης μετά από τις ταραχές και άρα εμείς δρούμε σε συνδυασμό με άλλους διεθνείς ε, φορείς. Επίσης σημαντικό και σωστό είναι βεβαίως ε, να υπάρχουν κάποια προαπαιτούμενα όπως η σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και βεβαίως δημοκρατία και κράτος δικαίου. Κατά την ε, χρήση αυτών των κονδυλίων θα πρέπει και οι δικές μας υπηρεσίες να συνεργαστούν με τις αρχές της Κυρκυζίας έτσι ώστε τα χρήματα αυτά να ξοδευτούν με τρόπο σωστό και αποτελεσματικό. Είναι λοιπόν για μένα σημαντικό αυτό γιατί βεβαίως η Κυργυζία δεν θα πρέπει να φτάσει να εξαρτάται από την βοήθειά μας, απλά θα πρέπει να τη βοηθήσουμε τώρα που αντιμετωπίζει κάποια διέξοδα. Η ίδια η κυβέρνηση της Κυργυζίας έχει δεσμευτεί για την σταθεροποίηση ε, των δημοκρατικών θεσμών και την προώθηση μιας διαδικασίας συμφιλίωσης. Όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν με τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να βοηθήσει εδώ πέρα, αλλά βεβαίως ε, δεν θα πρέπει να φοβηθεί και να ασκήσει ανοιχτή κριτική. Αλλά για να είμαστε αξιόπιστη δεν θα πρέπει να υποφέρει η Κυργυζία λόγω των εσωτερικών διαφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπουμε πως έχει τεράστια σημασία η Ασία για την Ευρώπη, γι' αυτό θεωρώ πως αυτή η μακροοικονομική συνδρομή είναι ένα θετικό μήνυμα για ολόκληρη την περιοχή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, ο κύριος Ρινάλντι. Αγαπητοί συνάδελφοι, Χωρίς να επαναλάβω τις ανησυχίες που ήδη εκφράστηκαν, είναι σαφές ότι αυτή η μακροοικονομική ε, συνδρομή είναι ύψης της σημασίας, όχι μας στα πλαίσια των εμπορικών σχέσεων, αλλά και της εξωτερικής μας πολιτικής. Το Κυργιστάν ε, ανταποκρίθηκε μετά την ανεξαρτησία του στις προκλήσεις μιας σκληρής μετάβασης ε, γνώρισε μεγάλους κλειδονισμούς. Τώρα ε, δυστυχώς βρίσκεται σε μια πτωτική πορεία, συμμετέχει στον ΠΟΕ, γνώρισε μεγάλες ε, περιφερειακές πολλούς περιφερειακούς κλειδονισμούς και αυτό έχει ένα αντίτιμο ιδιαίτερα σε μια χώρα με μεγάλη φτώχεια. Η συνδρομή ανταποκρίνεται σε ένα αίτημα ε, μεταρρυθμίσεων διαρθρωτικού χαρακτήρα και η Ρωσία και η Κίνα έχουν επενδύσει σε αυτή τη χώρα, γι' αυτό θα πρέπει και να είμαστε προσεκτικοί, ιδιαίτερα όσον αφορά την βιωσιμότητα κάθε μεταρρύθμισης σε μία φτωχή χώρα αλλά αξιοπρεπή και οι αρχές θα πρέπει να ξέρουν να προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και θα ήθελα να ε, πω και εγώ ότι ο Ασμάν Ισκάροφ ε, είχε γνωρίσει σοβαρές διακρίσεις. Ευχαριστώ ο κύριος Πέτερλε. Η κυριγησία τη μετασοβιετική περίοδο αντιμετώπισε το 2010 τρομερές συνέπειες. Τα γεγονότα αυτά επηρέασαν την οικονομία της χώρας αναπόφευκτα. Το 2010 οι πολίτες ψήφισαν για συνταματικές μεταρρυθμίσεις και η χώρα έχει, κινείται προς την κοινοβουλευτική δημοκρατία. Αυτή είναι σημαντική πρόκληση τόσο για την ίδια τη δημοκρατία όσο και για τις γειτονικές της τις χώρες. Προσωπικά το 2010 είχα την ευκαιρία να δω πόσο περίπλοκη ήταν η κατάσταση στη χώρα αυτή από πρώτο χέρι. Η Κυργυσία είναι μια χώρα η οποία αντιμετωπίζει δυσάρεστη μακροοικονομική κατάσταση και αυτή είναι μια πρόκληση για τις δημοκρατικές επιλογές της και είμαι πολύ ευτυχής που η Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ψήφισε για την συνδρομή αυτή και ελπίζω ότι θα την υποστηρίξουμε και εμείς. Ευχαριστώ κύριος Ανδρέας Μέλτσερ στη διαδικασία και Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κατάφερε να εδραιώσει την επιρροή της στην ε, πάρα πολύ σημαντική γεωστρατηγικά αυτή περιοχή και βεβαίως το ότι έπρεπε να παγώσει η Συμφωνία των 750 εκατομμυρίων δεν βοήθησε στην εμπιστοσύνη των χωρών αυτών. Η Κυργυζία είναι η μόνη χώρα της Κεντρικής Ασίας που πηγαίνει προς μία κατεύθυνση κοινοβουλευτικής δημοκρατίας αλλά ακόμα απέχει πάρα πολύ και βεβαίως πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τα βία γεγονότα του 2010 όπου είχαμε τραυματισμούς και βασανιστήρια. Οπότε παραμένουν ακόμα πολλά που πρέπει να γίνει βεβαίως. Το ζήτημα είναι το πώς θα προχωρήσουν οι πολιτικές μεταρρυθμίσεις και πώς θα γίνουν δεκτές από την κοινωνία. Ελπίζουμε πως η δική μας βοήθεια μαζί με τη βοήθεια της Ρωσίας θα βοηθήσει μια δημοκρατική εξέλιξη. Σας ευχαριστώ. Θέλει κάποιος άλλος να μιλήσει στη δικασία και Όχι, οπότε θα δώσω τον λόγο στον κύριο Επίτροπο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ορισμένα μέλη έθεσαν το ερώτημα γιατί χορηγούμε αυτή την μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή σε μια χώρα το Κυρικικιστάν που δεν ανήκει στην παραδοσιακή γειτονιά μας. Εγώ θα έλεγα, ωστόσο, ότι η δημοκρατία της Χιλισίας από στρατηγική άποψη ανήκει στην περιοχή μας, αλλά αυτό είναι ένα πολιτικό θέμα και μια πολιτική συζήτηση. Τα κριτήρια για την μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή που προβλέπεται σε ιδιάζουσες περιπτώσεις είναι μια δυνατότητα να ε, γίνουν επιχειρήσεις, να γίνουν προσπάθειες εκτός του κεντρικού κορμού των μακρο, της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής. Υποστήριξη για, το, ε, στη δημοκρατία, για τη δημοκρατία αυτή μια δημοκρατία εν το γεννάστε θεωρούμε ότι είναι σημαντική. Μιλάμε για ευάλωτη, για ευάλωτη ε, κοινοβουλευτική δημοκρατία. Το δέχομαι αυτό. Είναι και μια ευάλωτη χώρα, μια εύθραυστη χώρα την οποία πρέπει να βοηθήσουμε αν θέλουμε να προωθήσουμε και τη δημοκρατία. Η διατήρηση της οικονομικής σταθερότητας στη χώρα σε κρίσιμες περιόδους για να βοηθήσουμε τις δημοκρατικές αρχές και να αποφύγουμε την διεθνική βία η οποία θα διαχυθεί ενδεχομένως και στις τρίτες, ε, τρίτες χώρες, γειτονικές χώρες είναι ένας από τους στόχους μας. Είναι μια χώρα η Κυργυσία χωρίς φυσικούς πόρους και εξαρτάται εκ τούτου σημαντικά από το εμπόριο με τις γειτονικές της χώρες και πέρα από αυτό υπάρχουν και τα προβλήματα ε, μειονοτήτων όπως παραδείγματο χάρη με την ουσμπεκική μειονότητα. Χρειάζεται λοιπόν να παρέχουμε υποστήριξη, υποστήριξη στις χώρες που στηρίζονται σε δημοκρατικές αρχές με ατελή βεβαίω τρόπο. Δεν χρειάζεται να με πείσετε γι' αυτό, το γνωρίζω. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο. Το περιεχόμενο αυτής της απόφασης για την χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής. Μετά υπάρχει και η θεσμική πτυχή για το κατά πόσο μπορούμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου για τη διαδικασία που θα χρειαστεί να ακολουθήσουμε σε ό,τι αφορά και γι' αυτό εξαρτηθεί η ευθύνη μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Το θέμα είναι δεν πρέπει, όμως αυτό, ε, όμως να μην προωθηθεί αυτή η προσπάθεια. Γι' αυτό πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για να ξεπεράσουμε το αδιέξοδο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε. Τον τελευταίο λόγο έχει ο εισηγητής, ο κύριος Μαρέα. Ε, ε, Πρόεδρε, Υπάρχουν δύο λόγοι για την υποστήριξη αυτής της πρότασης της ε, Κομισιόν. Πρόκειται για μία επένδυση και μία δανειοδότηση μέσα στα πλαίσια των δημοκρατικών διεργασιών. Επίσης, η μακροοικονομική συνδρομή ε, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη ε, με τα ανθρώπινα δικαιώματα, διότι το άρθρο 5 αυτού του κανονισμού ε, μιλά για την καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε κατά πόσο πρέπει να απορρίψουμε αυτή τη μακροοικονομική σύνδρομη ή αντίθετα πρέπει να χορηγηθεί έτσι ώστε να πιέσουμε υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι η δεύτερη είναι η σωστή προσέγγιση, γι' αυτό και θα υποστηρίξω αυτή την πρόταση Επιτροπής και για την ε, μακροοικονομική σύνδρομη στο Κυρίσταν. Ευχαριστώ κύριε Σίγητα, κύριες και κύριοι. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση για αυτό το θέμα της ημερήσιας διάταξης. Η ψηφοφορία θα γίνει αύριο στις 12 η ώρα. Περνάμε τώρα.